Ε, η ε, πρόταση αυτή στο, στην, στην ιστοσελίδα. Επίσης, ε, η Επιτροπή Απασχόλησης έχει ενημερώσει για τέσσερις αλλαγές σε αντίστοιχα εγγραφά θα θεωρηθούν εγκεκριμένες εκτός και αν μέσα σε 24 ώρες δεν ζητηθεί συζήτηση και ψηφοφορία από 40 βουλευτές. Θα δημοσιευθούν λοιπόν τα κείμενα αυτά ε, και στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής. Θα ήθελα να σας πω ότι την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου